νομοθετικές πράξεις θα δημοσιευθούν αυτές στα πρακτικά. Και πάμε στον καθορισμό του προγράμματος αυτής της εβδομάδας, της συνόδου μας αυτής. Το τελικό σχέδιο προγράμματος υθετήθηκε στις 3 Μαρτίου από τη διάσκεψη των Προέδρων σύμφωνα με το άρθρο 137 του εσωτερικού κανονισμού και σας έχει δοθεί αυτό το σχέδιο του προγράμματος. Λοιπόν, καθημερινά θα καθορίζουμε την ημερήσια διάταξη. Τη Δευτέρα, λοιπόν, δεν έχουμε καμία αλλαγή όσον αφορά την αρχική μας πρόταση. Την Τρίτη, προσέξτε, την Τρίτη έχει γίνει μια αλλαγή. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων υιοθέτησε έκθεση του κυρίου Περόνιου όσον αφορά την άρση ασυλίας του κυρίου Έρμαρ Μπρόκ σύμφωνα με τις πολιτικές ομάδες και δυνάμει του άρθρου 138 αυτή η έκθεση θα συμπεριληφθεί στην ψηφοφορία αύριο. Είναι η κανονική συνηθισμένη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 138 του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την Τετάρτη και την Πέμπτη δεν έχουμε κάποιες προτάσεις για κάποιες αλλαγές σε σχέση με το πρωταθέν πρόγραμμα, οπότε μπορούμε να θεωρήσουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα ως εγκεκριμένο και μπορούμε να προχωρήσουμε στην πρώτη έκθεση. Συντάκτης είναι η κυρία Άννη Ποδηματά, η συνάδελφός μας, και ενωτόμα χρηματοδότηση σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κύριος Οντί κάτι θέλει να πει, έχετε το λόγο. Θα ήθελα να μιλήσω, ο Οντί, θα ήθελα να μιλήσω δυνάμει το άρθρο 16 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτή την εβδομάδα, κατόπιν πρωτοβουλίας του αρχηγού του κράτους, το οποίο νίκο του Νικολά Σαρκοζή, που ζητά ε, ε, να γίνει έκτακτο Συμβούλιο Ευρωπαϊκό την Παρασκευή να συνεδριάσει ήθιστε την εφαρμογή των συνθήκων το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων να προετοιμάζει τι συνεδριάσει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν είδαμε στην ημερήσια διάταξη αυτή τη εβδομάδα κάποια συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων την προετοιμασία τη εκτάκτου αυτή συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τη στιγμή μάλιστα που μεγάλα δημοκρατικά κινήμα και γονότα οι ευρωπαϊκοί λαοί θα πρέπει να συμμετέχουν μαζί με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων όσον αφορά τις ευρωπαϊκές τοποθετήσεις, όσον αφορά τα μεγάλα ευρωπαϊκά αυτά θέματα. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας αυτά. Και τώρα θα σας δώσω γραπτός απάντηση σε αυτό που μου είπατε. Και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε και να πάμε στην έκθεση.